με ονομαστική κλίση. I would now... Madam Geminas, yes? Yes. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να επωφελθώ που είμαστε όλοι εδώ για να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η μέρα που θυμόμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας ε, που συμπίπτει με τις 11 Μαρτίου όπου στην Μαδρίτη δεχτήκαμε αυτά τα τρομερά τρομοκρατικά χτυπήματα. Να πω με δύο λόγια ότι η τρομοκρατία ε, σκοτώνει ένα για να τρομοκρατήσει όλους τους υπόλοιπους και οποιοδήποτε από εμά μπορεί να γίνει θύμα τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό το σχόλιο. Ο κύριος Φιρέντσε, διαδικαστικό. Κυρία, μάλλον, συγγνώμη. Κυρία Φιρέντζε, διαδικαστικό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να επικληθώ τον κανονισμό σχετικά με ρατσιστική συμπεριφορά ενός ευρωβουλευτή του κοινοβουλίου μας, ο οποίος τους ε, Ρωμά τους ε, αποκάλεσε σε μια τηλεπτική εκπομπή ως μίασμα της ε, κοινωνίας και καλό τον, την πρόεδρο της αίθουσα να λάβει μέτρα έναντι του κ. Μπονάνο, ο οποίος προέβησε αυτή τη δήλωση. Could, could, could I please... Could I clarify for the... Παρακαλώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω. Θα ήθελα να διευκρινίσω. Okay, okay. Mr. Golnish, would you... Κύριε Γκόλνης, παρακαλώ, καθίστε, καθίστε κάτω, γιατί έχω να κάνω μία δήλωση και θα παρακαλούσα να ακούσετε με σεβασμό. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο σχόλιο τη κυρία Χιμένε, θα ήθελα να πω ότι ήδη έχει γίνει ανακοίνωση σχετική από τον πρόεδρο. Και δεν υπάρχει σχετική εντολή για δηλώσει ε, πέραν ε, της Ολομέλειας. Ε, αυτή η αυτή, αυτό, αυτό το σχόλιο για τους Ρωμά δεν έγινε στα πλαίσια της, ε, των κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Γι' αυτό δεν έχει σχετική αρμοδιότητα ο Πρόεδρος. Okay. Mr. could I, could I ask you, please... Κύριε Γκόλνης, παρακαλώ. Λίγη προσοχή για ένα λεπτό. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες να συνεννοηθούν μαζί σας και να διευκρινίσουν το κατά πόσο ήταν διαδικαστικό το σχόλιο σας. Στο μεταξύ θα περάσουμε στις ψηφοφορίες μέχρι ότου διευκρινιστεί το θέμα. Και παρακαλώ σεβασμός στην Ολομέλεια. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση, έκθεση Ντούντα για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Μαυροβούνιο. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση Ντούντα για τις δασμολογικές ποσοστώσεις ε, σε γεωργικά προϊόντα και άλλα υπολείμματα. Μία ψήφος με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση του κυρίου Ντούντα και πάλι με θέμα την εισαγωγή στην Ένωση Γεωργικών Προϊόντων Προέλευσης Τουρκίας. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτή. Επόμενη έκθεση Ντούντα. Και πάλι αφορά γεωρικά προϊόντα προέλευσης Τουρκίας. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Γκαμπριέλ Μάτο για την αλία στη Μεσόγειο με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση της κυρίας Ρέγνερ. Έτηση άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Ζαγοράκη. Διανατάσσεως της χειρός. Παρακαλώ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Ντούντα, πάλι δυνατά στις χειρός, πάλι η ασυλία, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Έκθεση Φερνάντες. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016. Πρώτη τροπολογία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η πρώτη τροπολογία. Τροπολογία 8. Διανατάσσου της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται. Επόμενη τροπολογία, η 9, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω ότι ήταν σαφή η διαφορά. Τροπολογία 11. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 14. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 4. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι λήξη. Απορρίπτεται. τραπολογία 30 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται τροπολογία 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση Φερνάντες. Περνάμε στην έκθεση Πυρίνσκι. Συγχαρητήρια στον εισηγητή τον προηγούμενο. Με θέμα την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος Άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3. Ψηφίσατε όλοι. Λέξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1 άρχεται ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά τη γνώμη μου ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Αν θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 2, κάνει μία αντίρρηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφίζετε όλοι λίγοι απορρίπτεται τροπολογία 54 υπέρ συγγνώμη παράγραφος 54 υπέρ κατά εποχές. Ας το επιβεβαιώσουμε. Παράγραφος 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 12. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. λήξη. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. εγκρίνεται. Περνάμε στο, στην έκθεση πρόοδου του 2014 για το Μαυροβούνιο. Ξεκινάμε με τροπολογία 1 με ανάταση της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Ας το επιβεβαιώσουμε. Ψηφίζουμε ονομαστικά για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Συγγνώμη, καταπίπτει. Περνάμε στην τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Επιβεβαιώνουμε την 2. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ψηφοφορία για την έκθεση πρώτου 2014 για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, Παράγραφο 1. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9 υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονική βεβαίωση για την παράγραφο 9 άρχεται λίγη απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην επόμενη έκθεση, έκθεση πρόοδου για τη Σερβία. Ξεκινάμε με τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επιβεβαιώσουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε συνολικά για το ψήφισμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην ψηφοφορία για το κοσυφοπέδιο τροπολογία 3 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Συγγνώμη, ζητήσατε ηλεκτρονική επιβεβαίωση για την 9. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την τροπολογία 9. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Ε, κάναμε λάθος το νούμερο. Για ποιο, για την τροπολογία 9 μιλάτε. Δεν έχει αποσυρθεί σύμφωνα με, με το δικό μου κατάλογο. Η τροπολογία 9 είχε αποσυρθεί αλλά επανακατατέθηκε και γι' αυτό και ψηφίσαμε επί αυτής. Και την απορρίψαμε. Τροπολογία 4. Εντάξει, διευκρινίστηκε. Ωραία, διανατάσσεως της χειρός. Ε, ποιος είναι υπέρ της 4. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για όλο το κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Ροζάτη. Ξεκινάμε με την τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για όλο το κείμενο άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην ε, έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του κυρίου Γκουτιέρεθ Πριέτο. Παράφος 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 3. Σε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Παράγραφος, ε, συγγνώμη, τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε Παράγραφος 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16 υπέρ. Για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράφος 17 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράφος 24 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Άρχεται η ψηφοφορία την 24. Παράγραφος 24. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα. Έναρξη, πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Λήξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με πολύ μικρή διαφορά. πράγμα 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 44 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Απορρίπτεται. Παράγραφος 47 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 49. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Παράφος 50 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 50. Έναρξη. Λήξη. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 54 σε δύο τμήματα. Όχι, συγγνώμη λέει Πρόεδρος, 52. 52 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 έχει αποσυρθεί. Παράγραφος 56 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λεξή. Εγκρίθηκε. Πράγμα 65 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι λέξη εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίφθηκε. Παράγραφο 69. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 71. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 παράγραφος 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε ηλεκτρονική βεβαίωση την παράγραφο 74. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Πράγμα 75 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Δεύτερο, ε, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε. Επιβεβαίωση ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Παράγραφος 78 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9. Ονομαστική σοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίφθηκε. Ε, το ιδιωτική γνώμη νη. Ε, ονομαστική σοφορία. Έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας W. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Υιοθετήθηκε. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία έκθεση Γκάλ Πέλτς για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Παράγραφος 17, μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ωραία λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή ψηφίζουμε το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Δεκτό. Ευχαριστώ. Κατόπιν έχουμε την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στο διαδίκτυο. Παράγραφος 15 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παραγραφούς 16 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος 18. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό εκτιμώντας L υπέρ κατά αποχές δεκτό εκτιμώντας μη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό τελική ψηφοφορία ονομαστική άρχεται και πέρας τελείωσε ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι Συνάδελφοι, λίγη ησυχία παρακαλώ καθώς φεύγετε από την αίθουσα. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Κύριε Γκόλνης, ε, έχει διευκρινιστεί αυτό το οποίο θέλετε. Δεν εμπίπτει κανονικά στον κανονισμό, αλλά έχετε τον λόγο για να μιλήσετε επί της διαδικασίας. Έχετε τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Διαπιστώνω ότι δώσατε το λόγο για διαδικαστικά επιθεμάτων τα οποία ουδεμία σχέση είχαν με τον κανονισμό λειτουργίας μας, ε, ούτε καμία σχέση με την σημερινή συζήτηση και μάλιστα ε, στη μία περίπτωση ε, αμφισβητήθηκε ένας από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πέστε μου λοιπόν συγκεκριμένα πού βασίσατε την αποδοχή ε, του την αποδοχή αυτού του διαδικαστικού να σας πω λοιπόν το εξή. Όταν έφτασα στο Στρασβούργο, οι συνάδελφοί μου και οι βοηθοί με μεγάλη έκπληξη μάθαμε ότι μας έδειχνε με το δάχτυλο δημόσια ο πρόεδρος ε, Σούλτς ε, για διάφορα θέματα και ότι ζητούσε από την γαλλική δημοκρατία να μας διώξει πριν καν δοθεί απάντηση από την Όλαφ στην οποία είχε στείλει το αίτημά του και μάλιστα δεν καταδέχτηκε ούτε καν να μας ακούσει όσον αφορά αυτές τις κατηγορίες τις οποίες δημόσια είχε ε, αναφέρει. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγράφος 4 εδάφιο 2 δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο. Βάσει δε ε, του άρθρου 5 ε, πρέπει να σας πω ότι παραβίασε την υποχρέωσή του να μας ακούσει. Επίσης Βάσει βάση του 2 παράγραφος 4 παραβίασε το δικό μας δικαίωμα όσον αφορά την ε, ε, ε, αξιοπρέπειά μας και μάλιστα κατηγόρησε το σύνολο των ε, βοηθών και των βουλευτών. Θα πρέπει να ξεκινήσει από τους βουλευτές και τους βοηθούς του, των σοσιαλιστών ε, γιατί διαφορετικά τα πράγματα δεν θα είναι ισόνομα. 30 χρόνια είμαι βουλευτής και ποτέ δεν είδα ένα πρόεδρο κοινοβουλίου, έναν πρόεδρο συνελεύσεως ε, να φέρεται με τέτοιο κομματικό τρόπο. Ευχαριστώ.